So, colleagues, uh, we uh, begin again on our 9.40. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε 9.40, τώρα είναι 9.43. Λέει ο Πρόεδρος. Είναι εδώ όλοι οι συνάδελφοι για το επόμενο θέμα, οπότε περνάμε στην παρουσίαση της μελέτης για ένα συνολικό σύστημα προστασίας των μειονοτήτων. Είναι μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή μας βάσει του ερευνητικού προγράμματος της ΛΥΜΠΕ του 2017. Και η σημερινή παρουσίαση βέβαια έχει να κάνει και με την υπόλοιπη ημερήσια διάταξή μας που δουλεύουμε ε, για έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά τις μειονότητες, έτσι, που θα την εξετάσουμε στις 4 Ιουνίου, κάτι που έχει βέβαια πολύ μεγάλη σημασία και για μας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Λίνα Βοσλιούτε από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών που έχει συντάξει από κοινού με κάποιον άλλον την ε, μελέτη αυτή. Έχετε το χρόνο. 10-15 λεπτά παρακαλώ. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε και μας δώσετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ καταρχάς που ζητήσατε να καταρτιστεί αυτή η πολύ σημαντική και επίκαιρη ε, έκθεση, μελέτη και από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ είχαμε επίσης συνεργασία πολύ θετική. Ήταν ε, ε, ο Σέρχιο Καρέ Πέτρα Μπάρτ, Ελσπετ Κάιλτ και εγώ ήμασταν τέσσερι συντάκτε. Ομαδική δουλειά έγινε. Και βέβαια βασιστήκαμε και σε γνώση ειδικών για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Σε Βελίνα Ρουσίνοβα, Αλέγκρε για τι θρησκευτικέ μειονότητε. Μπάστιαν Ντάβιτ Βαντερβέλτεν για τι γλωσσικέ μειονότητε. Αυτοί ήταν οι ειδικοί που μα βοήθησαν. Ένα από τα συνθήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πρόγραμμα σήμερα ε, λέμε επίσης ε, είναι η ενότητα και η διαφορετικότητα. Πώς όμως θα τα προστατεύσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Έχουμε ε, συνολικούς ολοκληρωμένους μηχανισμούς προστασίας των μειονοτήτων αυτή τη στιγμή. Διότι είναι κάτι αναγκαίο. Ε, λόγω της ανόδου ξενοφοβίας, αντισημιτισμού, ε, αντιτσιγκάνικης αφήγησης και τάσεων. Τα είδαμε και στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και σε πρόσφατες εθνικές εκλογές αυτά τα φαινόμενα. Όταν οι μειονότητες αρχίσουν να είναι θύματα της δράσης ε, της πλειοψηφίας, αυτό δεν είναι θετικό. Και νομίζω ότι είναι ε, μια σημαντική συνεισφορά αυτή η μελέτη. 170 σελίδες βέβαια είναι μεγάλη, αλλά μεγάλο μέρος της είναι παραρτήματα. Και ο στόχος της είναι να μελετήσει τα διεθνή συστήματα, τη σημεία εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρακτικά ζητήματα που άπτονται των μειονοτήτων στην παρούσα φάση και καλύτερη διασύνδεση του ζητήματος αυτού με τον μηχανισμό για το κράτος ε, δικαίου και την καλύτερη ενσωμάτωση στο σύστημα κράτου δικαίου, ώστε να μπορούν να προστατεύονται οι ακόμα και όταν υποχωρεί ε, η κατάσταση κράτους δικαίου σε κάποια χώρα. Έχουμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Έχουμε ένα τρίγωνο δημοκρατία, θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου. Αυτές είναι οι τρεις γωνίες πρέπει να σταθεροποιηθούν και να παραμείνουν άθικτες ε, οι τρεις πλευρές του τριγώνου. Οι μειονότητες ε, είναι κάτι διτό για μας. Από τη μία ε, πρέπει να δούμε τα δικαιώματα μιας ομάδας για παράδειγμα. Γιατί υπάρχει μια ομάδα μπορεί να δουμε τα δικαιωματα μια διαφορετικές μια ομαδα γλωσσικές, πολιτιστικές ε, ανάγκες, θα πρέπει ε, αυτά τα δικαιώματα και ανάγκες της μειονότητας να γίνουν σεβαστά, αλλά υπάρχει και η ανάγκη μη διακριτικής μεταχείρισης που είναι κάτι πολύ βασικό. Η αρχή της μη διάκρισης είναι μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία λοιπόν είναι το κεντρικό σημείο. Πώς προστατεύουμε τις μειονότητες όταν υπάρχουν ε, διαρθρωτικές θεσμικές μορφές διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος τους πεδίο εφαρμογή μελέτε, εθνοτικέ, γλωσσικέ ε, και θρησκευτικέ μειονότητες. Στου τσιγκάνου εστιάσαμε. Νομίζουμε ότι πρέπει να δράσει η Ένωση πάνω σε αυτό και στον αντισημιτισμό. Και σε ό,τι αφορά τη σλαμοφοβία επίσης ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε εκτενώς. Έπειτα στραφήκαμε στα κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά και στη Σερβία που βρίσκεται υποκαθεστώς προένταξης. Επίσης ε, είδαμε και μια διατομεακή ε, προσέγγιση το κράτος δικαίου ή μάλλον Ε, είδαμε το καθεστώς ε, και τις δυνατότητες που έχουν οι μειονότητες για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Αυτό εξαρτάται το καθεστώς διαμονής, ε, αν έχουν καθεστώς νόμιμης διαμονής, αν είναι υπήκοοι κάποιου κράτους μέλους της Ένωσης ή αν είναι υπήκοοι του τρίτου κράτους και για μας υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάλογα με την κατηγορία. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τούτε άσυλο είναι μια νέα κατηγορία μειονότητας κοινωνία των πολιτών απάντησε σε μια ιντερνετική έρευνα και είπαν ότι υπάρχει μικρή δυνατότητα για αυτούς τους ανθρώπους να ασχίσουν τα δικαιώματά τους. Οι πιο παραδοσιακές τώρα προσεγγίσεις επίσης έχουν υπονομευθεί. Έχουμε μία μελέτη επιτόπη ε, βιβλιογραφική, 75 ε, απαντήσεις είχαμε από 11 κράτη και υπάρχει ένα focus group ε, για την ισότητα και το Equinet και οργανώσεις ε, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Συνεργάζονται με την ομάδα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και αυτοί έδωσαν πολύτιμες συνεισφορές. Με ένα πόρισμα σημαντικό ήταν ότι αν δεν υπάρχει προστασία των ε, μειονοτήτων και δεν υπάρχει κάποιο φόρουμ ή κάτι θεσμικό που να προστατεύει τις μειονότητες, αυτό δείχνει ότι υποβαθμίζεται το κράτος δικαίου. Είναι ένα πρώτο δείγμα. Εμείς λοιπόν Θέλησαμε να δούμε ακριβώς το πλαίσιο του κράτους δικαίου, πώς μπορεί να προωθηθεί μέσω του κράτους δικαίου ε, η προστασία των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή 8% του πληθυσμού ε, με υπόβαθρο από καταγωγή από μειονότητα και ένα μεγάλο ποσοστό είναι γλωσσικές μειονότητες. Και στο άρθρο 2 λέγεται ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και έχουμε και το χάρτη των πληθών δικαιωμάτων, το άρθρο 22. Τα κράτη δεσμεύονται να σεβαστούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και υπάρχουν και άρθρα για τη μη διάκριση. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τις ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σχετική οδηγία για τα μειονοτικά δικαιώματα. Ο ΑΣΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΙΕ είναι οι οργανισμοί που θεωρεί κανείς ότι πρέπει να παρασπίσουν κυρίως αυτά τα δικαιώματα. Όμως υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε σε τρίτους όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης για παράδειγμα για να μας επισημάνουν ότι κάτι κακό ε, συμβαίνει. Έχουμε και στα δικά μας νομικά συστήματα κάποιες διατάξεις. Παραδείγματος κανένα υπάρχει θεσμική διάκριση ε, σε βάρος των Ρωμά, των Τσιγκάνων. Αυτό υποβαθμίζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη δικαστική ε, και ποινική συνεργασία. Αν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των Ρώμα, αν δεν λαμβάνονται υπόψη επαρκώς στο δικαστικό σύστημα ή αν ε, είναι ένα μεγάλο τμήμα των εγκλήστων σε φυλακές. Αυτό έχει να κάνει με τα εθνικά συστήματα και η αμοιβαία εμπιστοσύνη εδώ είναι ένα πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να το ελέγξουμε. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και από αρκετέ ε, υποθέσει ε, ενώπιον του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βλέπουμε και κάτι ακόμη. Σε ό,τι την ένταξη των Ρωμά, κάνει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρετίζουμε τα σωστά βήματα, τα βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμως ότι είναι μόνο οικονομικά ή κοινωνικά δικαιώματα το πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν και τα θεσμικά μοτίβα και πρότυπα διάκριση που πρέπει να μας απασχολήσουν. Επομένως, αυτό το οποίο υποστηρίζουμε στη μελέτη μας είναι ότι στη νέα περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα για την εθνική ένταξη των και την καταπολέμηση ε, της διάκρισης κατά των Αθήγανων. Η Εκπρόσωπ των Ρώμα θα μπορούσαν να ε, προσβάλλουν, να αμφισβητήσουν αυτές τις, ε, να καταδείξουν αυτές τις μορφές ε, διακριτικής μεταχείρισης και συμπεριφοράς. Επίσης, ότι τη χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία και των πολιτών. Ποιος εκπροσωπεί τελικά τις μειονότητες. Αυτό είναι ένα είδος πεδίου μάχης σε εθνικό επίπεδο. Συνήθω δεν είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν, που εκπροσωπούν τι μενότητε, αλλά αυτοί που έχουν καλύτερε διασυνδέσεις με αυτού που βρίσκονται σε θέση ισχύω. Επίση, τι άλλο ε, διαπιστώσαμε. Πόσο σημαντική είναι η ανεξαρτησία των ε, αρμόδιων για την ισότητα. Ένα από τα βασικά πρακτικά ζητήματα και πρακτική πρόκληση που μελετήσαμε και το βλέπετε ξεκάθαρα στα παραρτήματα είναι η μη συμμόρφωση σε διάφορους διεθνείς μηχανισμούς όπως το UPR για παράδειγμα. Επιτροπή εκρίζωσης ε, φιλετικής διάκρισης, Επιτροπή κατά της ε, διακριτής μεταχείρισης σε βάση των γυναικών και βλέπουμε ένα επαναληπτικό μοτίβο μη ε, με τους διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς και πρότυπα. Η ομάδα αυτή που σας είπα πριν, το Focus Group, διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποια κόποση στις κυβερνήσεις ε, ό,τι αφορά τη συμμόρφωση και έτσι κάπως τυποποιούνται αυτές οι καταστάσεις μη συμμόρφωσης και προτύπων ε, διεκτικής μεταχείρισης. Και αυτό το είδαμε και στις 11 χώρες που μελετήσαμε στη έρευνα. Uh, one, uh, one of the Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι συχνά στο επίκεντρο των εθνικών και περιφερικών μηχανισμών υπάρχει το θέμα της πολιτικής βούλησης ε, από πλευράς κρατικών φορέων. Υπάρχει ένας διαγωνισμός του ποιος θα είναι αυτός που θα πρωταγωνιστήσει στα θέματα προστασίας. Ε, αλλά πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα και δεν υπάρχει και παρκής έλεγχος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε εκεί να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο. Άλλα ζητήματα είναι. Η μη επικαιροποίηση ή η μη επικύρωση κάποιων συμβάσεων ή συνθήκων και πρέπει να δούμε ποια είναι τα κρατημέλη που δεν έχουν επικυρώσει, που δεν έχουν κυρώσει ποιε συμβάσει και ποιες διεθνείς ε, πράξει. Πανέρχομαι στο κράτος δικαίου. Τρία σενάρια. Για τα κρατημέλη. Να υπάρχουν ανέπαφα τα δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά οι εθνικοί μηχανισμοί επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεύτερο σενάριο είναι να υπάρχει θεσμική διάκριση ή ρατσισμό σε βάρος μειονοτήτων, αλλά λύνονται με την παρέμβαση των εθνών μηχανισμών. Και τρίτο σενάριο είναι το λεγόμενο institutional capture, όπου εκεί δεν μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα. Βλέποντας, λοιπόν υπόψη, έχοντας υπόψη του μηχανισμού αυτού του κράτου δικαίου, καλό θα ήταν να υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή για να δει τη συστηματικότητα, τη σοβαρότητα των παραβάσεων σε βάρος ευάλωτων ομάδων θα μπορούσε να συλλέξει στοιχεία για επίμονους κινδύνους και θα μπορούσε και να παρεμβαίνει πριν τα πράγματα περάσουν ε, στο τρίτο σενάριο που θα είναι αργά πια δηλαδή. Δείκτες τώρα για τη συστηματικότητα Το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ε, πλούσιο υλικό. Θα μπορούσαν να μελετηθούν κάποιες πιλωτικές περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε επίσης να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των ε, δικαστικών αποφάσεων και τα μέτρα δυνάμει του κανόνα 39. Προσωρινά μέτρα. Και ο χάρτης των πλέον δικαιωμάτων μπορούσε να είναι ένας νόμος κατά κάποιο τρόπο, ένα Bill of Rights. Να μην περιορίζεται η δράση της Ένωσης μόνο στο επικράτε της Ένωσης ή στους ενωσιακούς θεσμούς, αλλά να υπάρχει μια ευρύτερη δυνατότητα. Άρθρο 51 λοιπόν, το χάρτη των δικαιωμάτων, αυτό το άρθρο πρέπει να ε, αναβαθμιστεί, να διευρυνθεί το επίδιο εφαρμογή του. Και νομίζουμε επίση ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν ομαδοποιήσεις διαφόρων διαδικασιών παραβάση για να φανεί καλύτερα πώς παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι δεν αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρεμβάσει τρίτων θα μπορούσαν να έχουν σημασία όταν έχουμε κλίματα μίσου. και διακριτική μεταχείριση. αμίκου κούριε και δυνατότητα δρομολόγηση τέτοιων διαδικασιών ή άλλων διεθνών μηχανισμών. Μέτρα προσωρινά ή πάγωμα, μέτρα παγώματος, freezing, θα μπορούσαν να είναι επίσης αποτελεσματικά ώστε τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να δράσουν κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχουν κατατεθεί πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις από το κοινοβούλιο σας στον τομέα της ανεξαρτησίας ε, της κοινωνίας των πολιτών και της χρηματοδότησης ή ε, Balus Fund ερεσιμότητα, πρόταση για ένα νέο ταμείο ε, διαφορών, επίλυσης δικαστικών διαφορών κτλ. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ώστε να απολαμβάνουν ε, ίδιων ή παρόμοιων ε, δικαιωμάτων με τους άλλους ε, υπηκόους των χώρων που διαμένουν. Ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολλοί βουλευτές παρόντες. Εν πάση περιπτώσει... Όσον αφορά την ε, έκθεση του 2014, πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που ο Σέρζιο Καρέρα έχει ε, εμπλακεί γιατί πράγματι πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερος περίπλοκο και σοβαρό. Ιδιαίτερα σοβαρό και περίπλοκο. Ακόμα και ο ορισμός των ε, μειονοτήτων είναι ε, ζήτημα ε, και προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα το 2004 με τις ε, διευρύνσεις. Υπάρχει βέβαια και η οδηγία για την ποιότητα και, οδηγία, και άλλες οδηγίες οι οποίες είναι σχετικές με το θέμα και μπορεί κανείς να κατανοήσει ποια είναι η ιδέα που σχετίζεται με τις μειονότητες. CE and Council and so on makes E ε, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια, αλλά ιδιαίτερα περίπλοκη. Και το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η πολιτική και η στάση της είναι σημαντική. Ε, υπάρχουν οδηγίες σχετικές με το θέμα, οι οποίες όμως ε, δεν αντιμετωπίζουν πλήρως το θέμα. Κοιτάξτε, Βεβαίω εδώ αυτή η έκθεση έχει συγγραφεί σε σχέση με την έκθεση ίδιας πρωτοβουλία. Αλλά ελπίζω ότι πραγματικά θα την χρησιμοποιήσει ο κόσμος την έκθεση αυτή, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα. Στην περίπτωση της κυρίας Γκίλτ ε, είχαμε δικηγόρους ε, που προσπαθούν να βρουν μια λύση στο θέμα. Το ζήτημα είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξέρουν τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για αυτούς. Έχουν προταθεί ε, πάνελ αξιολόγησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί συνήθως η διαδικασία είναι δύσκολη για τις ε, μειονότητες. Είναι, μιλάμε για μειονότητες οι οποίες περνάνε από δύσκολες διαδικασίες, διαδικασίες ε, διακριτικής μεταχείρισης, ε, μη χρήση των μηχανισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη. Επομένως η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί προσπαθεί να βρει που ακριβώς εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιο τρόπο στα θέματα αυτά. Είναι αξιόλογη η εργασία. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Γιατί υπάρχει και ένα διεθνές δικαϊκό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά συστήνω στους συναδέλφους να, το, να διαβάσουν την έκθεση αυτή δεν είναι απλώς έτσι ένα καλογραμμένο κείμενο, ε, ε, περιλαμβάνει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι να υποβάλουν ερώτηση ε, όσον αφορά αυτή την έκθεση. Όχι, δεν ξέρω. Παρακαλώ. Κανείς. Ή εγώ έχω μια ερώτηση. Σχετικά με τις οδηγίες και τις μειονότητες. Φαντάζομαι Πώς ορίζετε εσείς ε, τις, ε, ε, τις μειονότητες, τι σημαίνει μειονότητα, ποια, αισθάνεστε ότι έχει αλλάξει αυτή, αυτός ο ορισμός και η κατάσταση τα με τον χρόνο, γλωσσικές μειονότητες κλπ. Πώς ορίζετε τις ομάδες οι οποίες υφίστανται διακριτική μεταχείριση πώς μπορούν να μπουν, ε, ε, να ταιριάξουν με, με, αυτήν την, με αυτούς τους ορισμούς ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αν ήμουν ο Ευρωπαίος πολίτης που και υφιστάμουν πιέσεις τι θα μπορούσα να προσδοκώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιο τρόπο θα μπορούσα να προσδοκώ να προστατευτώ, ε, με μια οδηγία, με κάποιον άλλο τρόπο. Εάν ορίσω τον εαυτό μου ως ε, μέλος μειονότητας που υφίσταται ε, διακριτική μεταχείριση και που χρήζει προστασίας. Ίσως βέβαια αν διαβάσουμε προσεκτικά όλη αυτή την έκθεση να καταλάβουμε τι γίνεται. Αν είσαι ας πούμε στην, ε, αν ανήκει στη μειονότητα Ρωμά, τι μπορείς να περιμένεις ε, από το νομικό σύστημα της ε, χώρας σου και από τη στιγμή που υπάρχει το νομικό σύστημα της χώρας σου, πώς, τι μπορείς να περιμένεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι έχει υπάρξει πρόοδος στο θέμα αυτό και στον τομέα αυτό, αλλά μήπως μπορείτε εσείς να μας πείτε κάτι παραπάνω. Έχουν προκύψει άλλωστε και οι σχετικές οδηγίες, ε, πρόκειται για ε, την οριζόντια οδηγία και πού αυτή μπορεί να ενταχθεί στο συνολικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ γιατί και για τα καλά σας λόγια και για την ερώτηση. Στην έρευνα, στη μελέτη αναγνωρίζουμε ότι όσον αφορά τους ορισμούς προς ώρας, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών να ορίσουν ποιες είναι οι μειονότητες και ποιοι ανήκουν σε, αυτούς, σε αυτές. Έχει ένα πλαίσιο το Συμβούλιο της Ευρώπης βεβαίως για τις μειονότητες που καθορίζει κάποια πλαίσια πέραν των οποίων δεν μπορούν ε, να πάνε τα κράτη-μέλη. Το ζήτημα δεν είναι όμως τόσο πολύ ζήτημα ορισμού και ποιες είναι οι μειονότητες, αλλά όταν ε, μιλάμε ε, για συστημική, θεσμική διακριτική μεταχείριση, τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Εκεί αναγνωρίζουμε ότι στην περίπτωση των Ρωμά πολλά έχουν γίνει μέσω του soft law και μέσω ε, συγκεκριμένων μέτρων και επομένως έχει κατά κάποιο τρόπο ξεπεραστεί η ανάγκη για, συγκεκριμένη, για συγκεκριμένο ορισμό. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν αυτά τα μέτρα μέσω των οποίων ε, ε, και οι μετακινούμενοι Ρωμά ε, και οι Ρωμά που είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αισθάνονται προστασία και πραγματικά θα έχουν την προστασία που χρειάζονται. Το 2010 είχαμε ας πούμε πολλές αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ε, ε, βίαιες απομάκρυνσης ε, Αθηγάνων Ρωμά στην Γαλλία. Υπάρχουν και οι εθνικές στρατηγικές σε των Ρωμά και νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποφύγουμε συγκεκριμένες στοχευμένες θεσμικές διακριτικές μεταχειρήσεις απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες. Όσον αφορά την ερώτησή σας πώς μπορεί να προστατέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με καλύτερο τρόπο τα μεμονωμένα άτομα, εάν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, πιστεύω ότι υπάρχει δυναμικό ε, για οριζόντια οδηγία. Αυτό είναι κάτι που εκρεμεί ακόμη. Οπωσδήποτε σε επίπεδο ατόμου θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ε, ε, δυνατότητες ατομικής ε, προστασίας, όπως προστατεύονται και άλλες εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. Αυτή τη στιγμή μονάχα η οδηγία Ρέιζε δίνει κάποια μεγαλύτερη δυνατότητα προστασίας σε ευρύτερα πεδία της ζωής και η οδηγία για την ισότητα ε, επίσης ε, καλύπτει κάποιες ε, ανάγκες προστασίας αλλά κυρίως στον εργασιακό χώρο. Υπάρχουν συστημικές, συστημικά επίπεδα, θεσμικά επίπεδα διακριτικής μεταχείρισης και εκεί υπερισχύει αυτή η, αυτή η αρχή της πλειοψηφίας που ανέφερα προηγουμένως λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει και κάποια εξωτερική ε, ε, παρακολούθηση ε, και εν πάση περιπτώσει εμείς θέλουμε το κράτος δικαίου να υπερισχύσει εντός του συστήματος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως έλεγα και προηγουμένως, πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, ουσιοδέστατο και σχετίζεται με την έκθεση ίδια πρωτοβουλίας ε, και με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειονοτήτων θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και το ΣΕΠΣΕ για την ε, εργασία του. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε νομίζω. Ε. Περνάμε στα σημεία 5, 6, 7 και 8 και 9 και 10. 11 και 12. Όλα αυτά τα σημεία αφορούν εκθέσεις, συστάσεις μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αποφάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση έναρξης διαπραγματεύσεων σχετικά με ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων ε, μεταξύ Europol και αρμοδίων ε, αρχών διαφόρων χωρών. 25 Απριλίου μας παρουσίασε η Επιτροπή της προτάσει. Πρόκειται για την Αλγερία, το Ισραήλ, το Ισραήλ την, την την Τουρκία, ε, η Ορδανία. Πρέπει σύντομα να ολοκληρώσει το Κοινοβούλιο για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα με τις χώρες αυτές. η Επιτροπή ενέκρινε τη σύστασή της στις 20 Δεκεμβρίου του 2017. Εγώ είμαι ο εισηγητής. Τι να σας εξηγήσω. Ακούστε με, παρακολουθήστε με λίγο. Το Συμβούλιο λοιπόν θέλει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ε, το Κοινοβούλιο στο τέλος των διαπραγματεύσεων δίνει τη σύμφωνη γνώμη του. Πρέπει να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή αλλά και τις ενδιαφερόμενες χώρες όσον αφορά τις αρχές, τους περιορισμούς και τα λοιπά των ε, διαπραγματεύσεων. Όπως τα έχετε διαβάσει, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει βέβαια, αν το διαβάσατε, λέει ότι η εντολή διαπραγματεύσεων πρέπει να σημειώνει τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι κάτι πολύ βασικό για μας και θέλουμε να υλοποιούνται τα δικαιώματα αυτά και να προστατεύονται των ε, ατόμων δηλαδή των οποίων τα δεδομένα μεταφέρονται. Δεν θα υπάρξει καμία αποδυνάμωση της προστασίας αυτής. Δεν θέλουμε να δεχτούμε καμία τέτοια αποδυνάμωση μέσω αυτής της απόφασης. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται η μεταφορά. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει και εκθέσεις αντικτύπου έτσι ώστε να ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια θέματα όπως είναι η παραπέρα επεξεργασία, η αποθήκευση, η αρχή της ιδιαιτερότητας και η απαγόρευση ανταλλαγής δεδομένων όταν πρόκειται για απάνθρωπη μεταχείριση είναι κίνδυνοι που για μας πρέπει να αποτελέσουν κόκκινες γραμμές. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τα είδη των εγκλημάτων και τον ορισμό τους. Οπότε, συνάδελφοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τις αρμόδιες αρχές για την προστασία δεδομένων, τις εθνικές αλλά και την ευρωπαϊκή. Βέβαια δεν ε, είναι όλα τα εποπτικά σώματα ίδια. Οπότε πρότασή μου είναι να συμπεριλάβουμε μια υποχρέωση για τις δύο πλευρές να καθορίζουν μια τέτοια αρχή η οποία θα μπορεί να αποφασίσει την πάυση, την αναστολή τη συμφωνίας σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση. Είναι σαφές ότι πρέπει η μεταφορά να γίνεται πάντα για το σκοπό για τον οποίο έχει ζητηθεί αρχικά. Και όταν πρόκειται για εθνική προέλευση, για πολιτικές απόψεις, θρησκευτικέ, ε, φιλοσοφικές ιδεολογίες κτλ. Ε, τέτοιες ε, Αν πρόκειται για τέτοιου σκοπού, δεν θα πρέπει να γίνεται αυτή η ανταλλαγή, εκτό αν υπάρχει κάποιο πολύ ιδιαίτερο λόγο. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί να τηρούνται οι προδιαγραφές μας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αποδυνάμωση αυτών δικαιωμάτων και είναι σαφές από την αρχή ότι εμεί θέλουμε να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με την χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα της υπευθυνότητας εφόσον υπάρξει παραβίαση της χάρτας αυτής είναι κάτι το οποίο πρέπει να τίθεται αμέσω και να αντιμετωπίζεται. Θα δώσω στους συναδελφούς τον λόγο. Έχουμε εδώ και εκπροσώπους της Επιτροπής του ETPS, το επόπτη προσωπικών δεδομένων δηλαδή, και οι συνάδελφοι εφόσον έχουν ερωτήσεις μπορούν να τις θέσουν. Ποιο θα πάρει το λόγο πρώτο. Ε, η κυρία Σίπελ. Παρακαλώ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ, σύντομα. Ναι, είναι μια συμφωνία για την οποία είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για όλες αυτές τις πολλές και διαφορετικές χώρες. Στην εισαγωγή σας αναφέρατε ήδη κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η κατάσταση σε αυτές τις χώρες που είναι στο κατάλογό μας βέβαια διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υπάρχει και διαφορετικό επίπεδο επεξεργασίας των δεδομένων και διαφορετικό επίπεδο ελέγχου που έχουμε εμείς το πώς γίνεται αυτή η επεξεργασία σε αυτές τις χώρες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή εμείς δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών δεν θέλουμε να δώσουμε σε χώρες για τις οποίες δεν έχουμε καμία εξασφάλιση για το τι θα τις κάνουν, τα κάνουν αυτά τα δεδομένα και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας μεταφοράς και που θα καταλήξουν επίσης αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό και είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Europol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε περισσότερες ε, λεπτομέρειες και απαντήσεις για την ε, τρέχουσα διαδικασία προκειμένου να δούμε τι άλλο θα πρέπει να γίνει. Οπότε, υπογραμμίζω και εγώ αυτό που είπατε και εσείς, ότι πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις με τα άλλα θεσμικά όργανα για να δούμε τι διακυδεύεται εδώ και πώς θα προχωρήσει η δουλειά τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλος. το Συμβούλιο, κύριος Ματσίσκη. Έχετε κάτι να πείτε σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Από τη δικιά μας την πλευρά, στο Συμβούλιο, εκπροσωπούμε εδώ την Προεδρία και είμαι και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας που συζητάει τις αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου. Είχαμε ήδη μέχρι τώρα έξι συναντήσεις όπου συζητάμε το σχέδιο απόφασης αυτό. Οι χώρες μέλη χρησιμοποίησαν κάθε ευκαιρία προκειμένου να επιμείνουν για το ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και ξεκάθαρες ρήτρες ασφάλειας και έλεγχος όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τη ελευθερία του ατόμου. Όπως είπατε κι εσείς, ήδη έχουμε τη γνωμοδότηση του EDPS, του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων, που προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να ε, συμπεριλάβουμε, να σωματώσουμε στο κείμενο. Στην επόμενη συνάντηση που είναι αύριο, ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω στο κείμενο να εγκριθεί μετά στην Κορεπέρ και σε επίπεδο Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, κύριε Σαμίτση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την σημαντική αυτή συνεισφορά σας. μας βοηθάτε όλους προκειμένου να προετοιμάσουμε την διαπραγματευτική διαδικασία. Ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με τις δικές σας ανησυχίες όσον αφορά την εξασφάλιση ότι οι μελλοντικές συμφωνίες αυτές θα διασφαλίζουν το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη χάρτα. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε κάνει πολλά για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι ρήτρε ασφαλείας αποτελούν πλήρως μέρος της οδηγίας που διαπραγματευόμαστε. Και όπως τόνισε και η Προεδρία μόλις πριν, ε, γίνονται συζητήσεις με τις χώρες μέλη για τα σχέδια όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της οδηγίας προκειμένου να ενισχυθεί το κείμενο και ελπίζω να διαπιστώσετε ότι οι οδηγίες και η απόφαση του Συμβουλίου που αναμένουμε να εγκρίνει σύντομα το Συμβούλιο προκειμένου να δώσει εντολή στην Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις, ότι θα αντικατοπτρίζει πλήρως λοιπόν, ελπίζουμε, αυτά τα οποία αναφέρετε και εσείς στο δικό σας σχέδιο έκθεσης. Όπως ήδη είπαμε, έτσι καλώς αντικατοπτρίζουν και πολλές από τις ανησυχίες του Ευρωπαίου Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων στη γνωμοδότησή του του Μαρτίου. Ένα σημείο θέλω να σχολιάσω. Η έκθεσή σας μιλάει για το ρόλο των εποπτικών αρχών στις τρίτες αυτές χώρες. Το να υπάρχει μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή φυσικά αποτελεί ακρογωνίο λίθο της προστασίας δεδομένων. Και αυτός είναι ένας στόχος για τον οποίο θα αγωνιστούμε. Όμως, το κατά πόσο μια τέτοια εποπτική αρχή έχει το δικαίωμα να πάψει να αναστείλει τη συμφωνία πιστεύουμε ότι πηγαίνει πιο μακριά από ένα σώμα, από μια αρχή προστασίας δεδομένων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των διαφόρων ρητρών προστασίας από την άλλη πλευρά. Εγώ θα έλεγα θα ήταν καλύτερα να υπάρχουν διατάξεις μέσα στην οδηγία που να μιλούν για μηχανισμούς εποπτικούς και για μια περιοδική αξιολόγηση ε, των συμφωνιών. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, Πρόεδρε, να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστω θα έρθει ξανά και ξανά στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. EDPS, Δερόφσκι, από την Υπηρεσία του Ευρωπαίου Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, τα περισσότερα στοιχεία που περιλάμβανε η γνωμοδότηση του επόπτη προσωπικών δεδομένων έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο κειμένου της συμφωνίας οπό, της απόφασης. Οπότε πρέπει να σας πω ότι μας ικανοποιεί η έκθεση έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα και πολλά σημεία που περιλαμβάνει η έκθεση είναι βασικά για το μέλλον των συζητήσεων. Θα σταθώ σε τρία που είναι πολύ σημαντικά για τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πρώτο έχει να κάνει με τη μεταφορά δεδομένων. Στην ε, έκθεσή μας Μάλλον στην έκθεσή σας που παρουσιάζετε σήμερα υπάρχουν δύο σημεία που λένε ότι η μεταφορά αυτή μέσα στην ίδια χώρα θα πρέπει να γίνονται μόνο για τον ίδιο και αρχικό λόγο για τον οποίο ζητήθηκαν τα δεδομένα και ότι οποιαδήποτε μεταφορά σε άλλη χώρα δεν επιτρέπεται. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πολύ βασικά για οποιαδήποτε υλοποίηση συμφωνίας, οποιαδήποτε συμφωνία. Έχουμε θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Και ελπίζουμε ότι όντως θα τηρούνται οι ρήτρες ασφαλείας. Δεύτερον, η έκθεση ζητάει να πούμε ότι η Europol θα τηρήσει τους περιορισμούς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Συμφωνώ ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν ένα νομικό σύστημα προστασιαμένο όπως το Ισραήλ, ενώ υπάρχουν χώρες που δεν δίνουν τέτοιες πληροφορίες όπως η Αλγερία. Οπότε, ακόμα και σήμερα, ευχαρίστως να σας ενημερώσω για την κάθε μία από αυτές τις χώρες χωριστά, εφόσον το επιθυμείτε. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, αλλά εσείς θα μου πείτε που είσαστε νομοθέτες. Ευχαριστούμε κύριε Βιριόσκη. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις. Η προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών είναι 30 Μαΐου. και τον Ιούλιο θέλουμε να πάει το θέμα στην Ολομέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέρφους που πήραν τον λόγο. Πάλι είμαστε νωρίς, δεν ξέρω, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Σίπολ. Επόμενο σημείο για το Σίπολ. χρειαζόμαστε συναδέλφους που δεν είναι ακόμα εδώ παρόντες, οπότε θα διακόψουμε για μισή ώρα. Πάμε πιο γρήγορα σήμερα από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Οπότε σημείο 14 για τη ΣΥΠΟΛ στις 11 ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση να έρθουν οι αρμόδιοι νωρίτερα. Ωραία, ναι. 30 λεπτά διάλειμμα. Επιστρέψτε παρακαλώ. στις 11 παρα 5. 11 παρα 5 να είσαστε εδώ παρακαλώ. 25 λεπτά διάλειμμα για το σημείο 14. 10.55, thank you. 10... Sorry, is it strange that it's 10.55 instead of 11? Όχι 11 λοιπόν, 11 παρα 5, έτσι, 11 παρα 5.

κάποιο δρόμο

Colleagues, thank you for your patience. We can... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Είμαστε στο σημείο 14. Είχαμε πάει πολύ γρήγορα, έτσι, είχαμε προχωρήσει γρήγορα και γι' αυτό διακόψαμε μετά. Οπότε είμαστε τώρα στο σημείο 14 που είναι η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας της ΛΥΜΠΕ στην ε, στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για κατάρτιση όσον αφορά την συμμόρφωση στον νόμο. Πήγαμε εκεί 5 και 6 Απριλίου. Η κυρία Γκάλ είναι η συγγήτρια για αυτό το θέμα, δηλαδή είναι η συγγήτριά μας για τον κανονισμό ΣΕΠΟΛ, ήδη από το 14-15. Είναι και ο κύριος Μάμικινς εδώ. Πρώτα η κυρία Γκάλ και μετά ο κύριος Μάμεκίνς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρέπει να πω δύο λόγια λοιπόν για την αποστολή αυτή στη ΣΥΠΟΛ. Πήγαμε τον Απρίλιο. Την έκθεση μπορείτε να τη διαβάσετε έτσι και αλλιώς ό,τι είναι σημαντικό είναι στην έκθεση. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να υπογραμμίσω τα πιο σημαντικά μηνύματα από την επίσκεψη αυτή. Να πω αυτής εξ αρχής ότι είναι σπάνιο να έχουμε μία αποστολή όπου να αναγνωρίζετε το τι κάνουμε εμείς εδώ. Αυτό που μας είπε λοιπόν το προσωπικό της ΥΠΟΛ είναι ότι οι προτάσεις μας για αλλαγές, για την εντολή της ΣΥΠΟΛ είχαν έναν ε, αυτό αντίκτυπο στη δουλειά των ανθρώπων εκεί. Είναι ερευνητικό κέντρο κατάρτισης. Πολλές φορές δεν ξέρανε τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν, ενώ τώρα είπαν ότι νιώθουν πως πραγματικά ε, μπορούν να έχουν την κατάρτιση αυτή που χρειάζεται για θέματα ασφάλειας, για τη μετώπιση της τρομοκρατίας και ότι είναι σε θέση πια να διδάξουν αυτά ακριβώ που ζητάει ο κόσμος, έχουν εμπειρία για να βοηθήσουν αυτούς που δρούν επιτόπου. Και λένε ότι αυτό έγινε ακριβώς επειδή εμείς φροντίσαμε να αλλάξει εντολή. Άρα λοιπόν μα ευχαρίστησαν για αυτά που κάνει η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που για αυτούς ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, για να είμαι σύντομη. Στόχος της αντιπροσωπείας μας ήταν να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις ε, του έργου του ΣΥΠΟΛ βάσει του νέου νομικού πλαισίου μετά το 2016. Η αντιπροσωπεία μας, εγώ και ο κύριος Μάμικινς από τους σοσιαλιστές, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκτελεστικό διευθυντή, τον αναπληρωτή και άλλο προσωπικό ε, της ΣΥΠΟΛ. Και οργανώθηκε πραγματικά από τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ πάρα πολύ καλά επίσκεψη αυτή. Και φαίνεται αυτό και στην ε, έκθεση. Ήμασταν λοιπόν στην έδρα της ΣΥΠΟΛ. Μας ξενάγησαν οι γκρικές αρχές υπήρξε κάποια ανακαίνιση από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας οπότε τώρα έχουν ένα πολύ ωραίο κτίριο, μια πολύ καλή τοποθεσία δεν έχουν όμως αρκετό χώρο από ό,τι φαίνεται επειδή αναλαμβάνουν όλο και περισσότερα καθήκοντα και επειδή υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το έργο τους. Ο κύριος Ρούντερ, ο διευθυντής, είπε ότι μας μίλησε για την αλλαγή του ονόματος, έτσι, από σχολή, από ακαδημία που ήταν πριν, για να ανταποκρίνεται καλύτερο τίτλο στα πραγματικά καθήκοντα της ε, ΣΥΠΟΛ. Επίσης, η υπηρεσία έχει σαν στόχο όχι μόνο τη στήριξη και το συντονισμό, αλλά και την υλοποίηση της κατάρτισης και να φροντίσει για νέα εργαλεία και νέα προϊόντα εκμάθησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το 2017 λοιπόν στα πλαίσια ε, των γρήγορων αλλαγών στις πολιτικές προτεραιότητες ανέλαβε ε, πάρα πολλές πρωτοβουλίες, 150 εκπαιδευτικές, ακόμα και online, Για να καταλάβετε πώς ακριβώς δουλεύουν όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι το 2014 οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες ΣΥΠΟΛ ήταν κάπου 10.000 και το 2017 έχουμε 23.700 συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της ΣΥΠΟΛ και η έρευνα ικανοποίηση των πελατών δείχνει ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν και προσωπικό πλέον που βρίσκεται σε κανονική λειτουργία. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, αλλά είναι και η γνώση, η ενημέρωση που βοηθάει πάρα πολύ το προσωπικό που ασχολείται με τη συμμόρφωση των νόμων και αυτό τα λένε όλοι οι ειδικοί. Υπάρχει επίσης ένα κέντρο γνώσης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Υπάρχει ε, συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών, παρόλο βέβαια που τα διάφορα αστυνομικά σώματα βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα προετοιμασίες. Όμως με την κατάρτιση αυτή ευθυγραμμίζεται κάπως η κατάσταση. Υπάρχει και το θέμα ε, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Υπάρχει το θέμα του σοβαρού εγκλήματος και του διασυνοριακού εγκλήματος. Υπάρχει επίσης πειραματικό πρόγραμμα για εταιρική σχέση με την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Διδάσκουν δηλαδή και μεταφέρουν γνώση στο προσωπικό επιτόπου τι να κάνουν σε περίπτωση που έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση τρομοκρατίας. Επίσης, η πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι βασικό στο έργο της ΥΠΟΛ. Τονίστηκε από τον κύριο Σιρούντερ αλλά και από άλλους στο προσωπικό ότι έχουν όλο και μεγαλύτερο φόρτο εργασίας χωρίς όμως να έχουν περισσότερο προσωπικό αντίστοιχα. Αυτό υπόθηκε πολλές φορές στις συναντήσεις μας και υπογραμμίστηκε ξανά και ξανά στις συζητήσεις. Το επόμενο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να προσφέρει περισσότερα κονδύλια στο τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Και για να ολοκληρώσω. Εγώ προσωπικά εκτίμησα πάρα πολύ το έργο της ΥΠΕΛ και βάσει των αποτελεσμάτων και της φήμης που έχει αποκτήσει η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι η επιλογή μας εδώ να διατηρήσουμε ένα ειδικό σώμα για την κατάρτιση των όσων ασχολούνται με τις μόρφωσεις των νόμων είναι μια σωστή επιλογή. Να ξέρετε ότι πρέπει να αυξηθούν οι πόροι της ΣΥΠΟΛ, γιατί κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο έργο. Φαίνεται αυτό, ε, η εντολή και τα καθήκοντα ε, γίνονται όλο και περισσότερα, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα αύξηση στο προσωπικό, στους ανθρώπινους πόρους. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάμεκινς που ήταν μαζί μου στις συναντήσεις αυτές και με συνόδευσε στις συζητήσεις. Και ευχαριστώ και το προσωπικό της Λίμπε για το δικό του έργο και για την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιο συνάδελφος θα ήθελε να μιλήσει για τη ΣΥΠΟΛ. Αν όχι να ευχαριστήσω την κυρία Γκάλ και να επενθυμίσω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή μας να παρακολουθεί εκ του σύνεκη σε το έργο των ε, οργανισμών ε, και άλλων υπηρεσιών και βέβαια να τις επισκέπτεται και τακτικά, όπως προβλέπουν οι κανόνες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τις ψηφοφορίες στις 11 και 15, η ώρα είναι 11 και 6. Περιμένω να προσέλθουν και άλλοι συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά από τις 11 και 4 και μετά. Άρα δεν μιλάω μέχρι τις 11 και 15. Κλείνω το μικρόφωνο και σταματώ εδώ.

Παρακαλώ καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι για να ξεκινήσουμε με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και σας υπόσχομαι να μην καθυστερήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Μια ανακοίνωση την οποία έκανα και στην αρχή της ε, συντήρησης, επιτρέψτε μου να επαναλάβω. Ο συγητής ε, για τα περί πιστευτικότητα συζήτησε με τις ε, ομάδες και θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία των συμβαστικών τροπολογιών. Και λόγω προσέλευσης το θέμα αυτό ε, για τα θέματα προστασίας ιδιωτικότητας δεν θα ψηφιστεί στην σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων ότι αυτό θα ήταν το λογικό. Θα αναβληθεί η ψηφοφορία, θα γίνει όμως το συντομότερο δυνατόν σε μεταγενέστερο στάδιο και να περάσουμε στην επόμενη τώρα ψηφοφορία. Έκθεση τα σχέδια απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να καθίσετε. Παρακαλώ, ησύχω. Να ψηφίσουμε λοιπόν το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για την ε, θέση σε εφαρμογή των υπολείπων διατάξεων ε, του κοινοτικού και εκτιμένου για Βουλγαρία-Ρουμανία σε ό,τι αφορά το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Δεν είναι σωστό ο αριθμό αναφορά. F15α20 κάθετος 1-2007 Rev 1 είναι ο σωστός τίτλος. Ε, θέλετε να πείτε κάτι παρακαλώ εσείς. Ναι, είμαστε πολύ πιο κοντά στο Σέγγιν σήμερα. Μιλώ για Ρουμανία και Βουλγαρία που βλέπουν πλέον τις προειδοποίησεις ε, άλλων κρατών μελών για την άρνηση εισόδου ή εξόδου σε κάποια κράτη αλλά δεν βλέπουν τα άλλα κράτη της ε, προειδοποίησης ε, της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Τώρα, με την έκθεση που ψηφίζουμε, αυτές οι αλλαγές θα μπορούν να τις βλέπουν όλοι. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει συνεργασία σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο ε, που θα βελτιώσει τη συνεργασία μας στο επίπεδο του Σέγγεν. Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών φυσικά είναι κάτι καθοριστική σημασία για όλους μας. Εξού και τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους και να εισάγουν τα σωστά δεδομένα. Ωραία, να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Δεν υπάρχει καμία τροπολογία. να αποσυρθεί και θα ψηφίσουμε ονομαστικά το σύνολο τη έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. That is 34 votes for, one against and two abstentions. 34 ψήφοι υπέρ, μία κατά δύο αποχές ε, εγκρίνεται και συγχαίρουμε την κυρία Μακοβέ, την εισηγήτρια. Και περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία Ε, σύμφωνα με τα εξοπλισμένε πολιτικέ ομοσπονδίε των διπλωματικών συμφωνιών, χρηματοπιστή ή στον τομέα των ψηφιακών συνόρων των θεωρήσεων. Άρχιτη τη ψηφοφορία, τέρμα, πέρμα τη ψηφοφορία. 34 ψήφοι υπέρ, μία κατά τρει αποχέ. Και επόμενο. Συμφωνία με τι Ευρωπαϊκέ Ένωσε και τη Ισλανδία, διπλωματικό ανασυντόνιο χωματοδοσία των ανεξαρτητών και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Στέγη Ασφάλεια. Βίστησεν, γιατί Θέλετε το λόγο, κύριε Βίστησεν. Α, δεν είστε εδώ. Δεν είναι εδώ ο κύριο Βίστησεν. Πώ να πάρει το λόγο, δεν είναι. Παρόν. Εντάξει, εντάξει. Βιάζεστε, έχετε να πάρετε κανένα αεροπλάνο, τι γίνεται. Λοιπόν, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 33 ε, ψήφοι υπέρ, ε, μία κατά και μία αποχή. Έπειτα το επόμενο θέμα είναι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ε, την ε, επιλογή του υποψηφίου για την Επιτροπή Επιλογής για το Διορισμό του Ευρωπαϊκού Γενικού Εισαγγελέα, ηλεκτρονικά και ε, μυστική θα είναι η ψηφοφορία που ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 34 ψήφοι υπέρ 3 κατά μια αποχή για τον κύριο Μούρα λοιπόν ο οποίος ορίζεται μέλος της Επιτροπής Επιλογής. Ολοκληρώσαμε 4 Ιουνίου, 3 το μεσημέρι, επόμενη συνεδρίαση. Γεια σας.